Τώρα κύριε και κύριοι, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξης, που είναι σημείο του κυρίου Μαρινέσκου για τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης αφορά όλα τα επίπεδα ζωής, όλα τα κράτη, ειδικά όταν μιλάμε για τα αυτοκίνητα. Όλα τα συστήματα είναι εξαρτημένα. Ε, έχουμε τέσσερις ε, δορυφόρους αυτή τη στιγμή και άλλοι 18 θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Το έγνος είναι το σύστημα το οποίο ενισχύει το μηχανισμό και θα εξασφαλίσει σημαντικές υπηρεσίες, θα καταστήσει δυνατό στα σήματα να ανταποκριθούν στις ανάγκες για, ανάγκη, στην ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία, παραδείγματο χάρη προσδιορισμό θέση, ακρίβεια κτλ. Οι μεταφορέ, η γεωργία, η ενέργεια χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα, τέτοια δορυφορικά συστήματα, και οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποφεληθούν από το Γαλιλαίο και το έγνο σε διάφορους τομείς. Παραδείγματο χάρη ε, αστυνομία, διαχείριση κρίσεων, ε, έκτακτες υπηρεσίες, διαχείριση των συνόρων κτλ. Η ανάπτυξη αυτών των δορυφορικών συστημάτων θα είναι υποφελής ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάπτυξη της επακόλουθης αγοράς και της ανάντη και της κατάντη δηλαδή αγοράς θα υπάρξουν ε, επιπτώσεις και για άλλους τομείς, θα δημιουργούν νέες θέσεις αποσχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματίες. Σε αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίες, το έγνος και το γαλιλαίος έχει ε, εξασφαλίσει μεγάλα κέρδη 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη οικονομική διαχείριση, γι' αυτό πρέπει να γίνει καλύτερο σχεδιασμό του προπολογισμού. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, την, με τις συμφωνίες για τους χερσαίους σταθμούς, τους ορφουρικούς σταθμούς, για την εκμετάλλευση των σημάτων έγνος ε, και με την διαχείριση των προγραμμάτων. Η Κομισιόν είπε ότι ένα εκατομμύριο ευρώ ε, κατέτος για τα 7 χρόνια από το 2014 μέχρι το 2020 είναι το νούμερο που μας είπε. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια ευέλικτη προσέγγιση, έτσι είπαμε στην Κομισιόν, ούτω ώστε η Κομισιόν να μπορεί να μεταφέρει κονδύλια από το ένα τομέα στον άλλο. Προς το παρόν, το 7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ εξαρτάται τους δορυφόρους, από αυτά τα συστήματα δηλαδή. Η υποστήριξη για τις εφαρμογές εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. 150 για την ε, τεχνολογία και άλλα 150 για την έρευνα και την ανάπτυξη. 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για την ανάπτυξη των εφαρμογών και το υπόλοιπο προβλέπεται να δοθεί από τον ορίζοντα 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει στον οργανισμό ευρωπαϊκού GNSS το ρόλο διαχείρισης του συστήματος. Θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο λοιπόν στο μέλλον και θέλουμε η Κομισιόν να ετοιμάσει ένα σχέδιο για να αναπτυχθεί αυτή η αγορά. Τελευταίο και σημαντικό, ο ρόλος καλής διακυβέρνησης που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη να δημιουργήσουμε στόχους και σαφή ρόλο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την Κομισιόν, για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκού GNSS, ESA, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο ε, και τις εθνικές, τους εθνικούς οργανισμούς, ούτως ώστε να υπάρξει σωστή εκμετάλλευση. Αυτοί οι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν και να είναι λειτουργικοί, μα, λειτουργική, συγγνώμη, μακροπρόθεσμα και ο καθένας να ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ταγιάννη. Έχετε το λόγο κύριε Ταγιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλος ιδιαίτερος και ιδίω τον κύριο Μαρινέσκου για τη δουλειά που έκανε πάνω σε αυτό το φάκελο. Όχι μόνο γιατί το Γαλιλαίος ήταν η πρώτη πρόταση τομεακή των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, ε, επί της οποίας ε, επετέχθη μια πολιτική συμφωνία, αλλά και γιατί το αποτέλεσμα, και κυρίως γιατί το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό, αυτή η συμφωνία μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειαζόμαστε θα δοθούν στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού στην ε, ανάπτυξη και χρήση του Γαλιλαίου και στις εφαρμογές του. Ευχαριστώ για τα σημαντικά αποτελέσματα που πετύχαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Το Γαλιλαίος έγινε μια πραγματικότητα τέσσερις ε, δορυφόροι είναι σε τροχιά και διάφοροι χερσαίοι σταθμοί, σταθμοί εδάφους δηλαδή υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Το, οι δοκιμέ που έχουν γίνει σε αυτούς τους τέσσερις δορυφόρους ε, δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε καλά. Από τα πειράματα που κάναμε τον Ιούλιο στην βάση του Φουκίνο με τους τέσσερις δορυφόρους ε, είδαμε ότι η θέση ο προσδιορισμός της θέσης χάρη στους τέσσερις ε, ε, δορυφόρους είναι πάρα πολύ ακριβής, ε, καλύτερη από τις τα αμερικανικά GPS. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα αυτά στο μέλλον θα λειτουργήσουν με θαυμάσιο τρόπο. αυτό δείχνει πραγματικά την ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα. Η ενεργοποίηση του προγράμματος συνεχίζεται, παρότι υπήρξε μια καθυστέρηση μερικών μηνών για την εκκίνηση και την τρομολόγηση των επόμενων δορυφόρων. Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι αισιόδοξο και είμαι πεπισμένο ότι πριν από την ολοκλήρωση της δικής μου θητείας ως Επιτρόπου για τη Βιομηχανία θα ε, είναι έτοιμη η πάροχη υπηρεσιών, δηλαδή οι πρώτες υπηρεσίες του Γαλιλαίου θα υπάρχουν ήδη από τον Οκτώβριο του 2014. Είναι σημαντικό αυτό για τους πολίτες μας και για τις ε, βιομηχανίες να μπορούν δηλαδή να υποφεληθούν το συντομότερο δυνατόν από τις ε, υπηρεσίες που προσφέρει το Γαλιλαίος. Το Γαλιλαίος είναι μια τρομακτική ευκαιρία για την ε, επανέναρξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός που συζητάμε σήμερα το βράδυ είναι ουσιαστικό βήμα για να εξασφαλίσουμε την συνέχεια του προγράμματος στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο. Όχι μόνο, σημαντικό όχι μόνο για οικονομικό, ως προς τους οικονομικούς όρους και ως ό,τι αφορά τη διαχείριση, την διακυβέρνηση του προγράμματος. Η Κομισιόν μεγάλη ικανοποίηση είπε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποστήριξαν πλέρια τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η διακυβέρνηση είναι μια σημαντική εξέλιξη στο οργανωτικό σχήμα του προγράμματος και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ε, εξορθολογισμού της χρήσης των υπάρχουσών υποδομών. Μέχρι μέσω μια νέα δομή, η Κομισιόν θα είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των, προγραμμάτων υπό τον πολιτικό έλεγχο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ τα διάφορα τεχνικά καθήκοντα για την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την υποδομή του συστήματος θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και στην, ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, GNSS. Το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα τμήμα του προπολογισμού που κινητοποιείται μέσω αυτού του ε, κανονισμού να δοθεί στη χρηματοδότηση ε, νέων οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει το έγνος και το Γαλιλαίος. Σε αυτό το πλαίσιο κρίσης που περνάει η Ευρώπη, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία, την οποία δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι, να μας φύγει μέσα από τα χέρια. Ζήτησα από τη Γενική Διεύθυνση να ε, εξετάσει όλες τις ε, εναλλακτικέ λύσεις και υπάρχει η ιδέα ε, ενός κειμένου, νομοθετικού κειμένου για τη χρήση του Γαλιλαίου. Θα ήθελα πριν κλείσω να σας πω ότι η Κομισιόν ξέρει πολύ καλά ότι τα 7 δισεκατομμύρια ε, για το πρόγραμμα για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο είναι ένα ανώτατο όριο. Δεν μπορούμε να το ξεπερνούμε, να το ξεπεράσουμε. Επομένως θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στο πρόγραμμα για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εμπλακούν ε, πολύ στα προγράμματα και θα υπάρχει μια αιτήσια έκθεση ε, των δικαιούχων για την εξέλιξη του προγράμματος. Η Κομισιόν θα συνεδριάζει τακτικά με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο εσωτερικό των ε, διαθεσμικών επιτροπών που υπάρχουν για το Γαλιλαίο, όπως έγινε ακριβώς και το Νοέμβριο όπου τα κοινωνικά, κοινοτικά θεσμικά όργανα ενημερώθηκαν για όλα όσα συμβαίνουν και για τα τεχνικά θέματα. Ε, ευχαριστώ όλους και τον επικεφαλής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Τέρχο. Συνεχίζουμε με την κυρία Καρβάλιο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την εξαιρετική του έκθεση. Με το πρόγραμμα Γαλιλαίο έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης πολύ πιο προηγμένο που εξασφαλίζει μια ακριβή, ένα ακριβή προσδιορισμό και αξιόπιστο προσδιορισμό θέσης. Πρόκειται για ένα εμβληματικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτει στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία θα είναι πρώτη που θα υποφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό το Γαλιλαίο συμβάλλει στη λειτουργία πολλών οικονομικών τομέων και δίνει σε επιχειρήσεις ε, και τους πολίτες άμεση πρόσβαση σε ένα σήμα πλοήγησης ε, μέσω δορυφόρου και μάλιστα ευρωπαϊκού. Είναι σημαντική η ευρωπαϊκή διάσταση και η προστιθέμενη αξία αυτού του σχεδίου. Γι' αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να τύχει της κατάλληλης χρηματοδότησης και γι' αυτό έδωσε 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ. Και τώρα για 1,5 λεπτό το λόγο η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μαρινέσκου, ο οποίος προετοίμασε μια θαυμάσια έκθεση και μας δίνει την ευκαιρία για εξαιρετικές συζητήσεις. πάντοτε στα μεγάλα σημαντικά θέματα εξαρτώμεθα από βασικά ζητήματα υποδομής ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή με το GPS. Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία των Αμερικανικών δορυφόρων και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό προσπαθούμε να πιέσουμε ώστε να έχουμε δικές μας ευρωπαϊκές δομές το Γαλιλαίο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πολύ σημαντική αρχή, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας από το αμερικανικό GPS. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επί πολλά χρόνια ε, είναι υπέρ μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ε, διαστήματος που θα είναι ανεξάρτητη από τις αμερικανικές υποδομές. Πάντοτε παλεύαμε υπέρ του Γκαλιλαίου, πάντοτε θέλαμε να έχει τη σωστή χρηματοδότηση στον Γαλιλαίο και νομίζω ότι πλησιάζουμε προς αυτό το στόχο ώστε να έχουμε μια βιομηχανία υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη που να έχει τη δυνατότητα να μας δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Είμαι αισιόδοξη και νομίζω ότι στο τέλος ε, με 27 δορυφόρους ε, σε τροχιά θα μπορέσουμε να έχουμε ε, την επιχειρησιακή ικανότητα που χρειάζεται τον Καλλιλέο. Ευχαριστώ. Μια γαλάζια κάρτα για σας. Τη δέχεστε κυρία Νίμπλε. Κυρία Νίμπλε. Ε, γαλάζια κάρτα από τον κύριο Γκασπάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφε Νίπλε, Είχε συζητηθεί πριν από λίγο καιρό αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να έχουμε τόσα χρήματα στη διάθεσή μας να χρησιμοποιούμε για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. ούτως ώστε να είναι ε, ένα ε, εγχείρημα που θα έχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην προσθέσουμε σκουπίδια στο διάστημα. Ευχαριστώ, συνάδελφε Κασπάρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα και βεβαίω και θέλω να το απαντήσω. Ε, όντως, τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε τη σκέψη μας και να εξελίσσουμε τα επιχειρηματά μας ε, και την επόμενη, στην επόμενη Ολομέλη το Δεκέμβριο ε, θα συζητηθεί ε, μια δική μου έκθεση για την πολιτική ανάπτυξη που άπτεται και αυτών των θεμάτων και νομίζω ότι πολλά τέτοια θέματα έχουν τεθεί προς συζήτηση και μια έκθεση του κυρίου Πρόντι για το Κοπέρνικους ούτως ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε με τα χρήματα των Ευρωπαίων Φορολογουμένων μια υποδομή που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσει πρόσβαση στι δικέ μα επιχειρήσει, στις μικρομεσαίες επιχειρήσει, και ούτω ώστε να μπορέσουν να, να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν και εδώ και πολλούς μήνες θα σκεφτόμαστε αυτά και ε, ακόμη στην τρέχουσα νομοθετική περίοδο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτριά μας είναι η κυρία Τσικάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. το γεγονός ότι έχουμε ε, ένα ανώτατο ποσό 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το έγνος και το Γαλιλαίο από το κοινοτικό προϋπολογισμό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 είναι σημαντικό γιατί η χρήση αυτών των συστημάτων δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα και οι υπηρεσίε που προσφέρουν το Γαλιλαίο και το έγνος είναι πολύ σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία μεγάλο αριθμό οικονομικών κλάδων όπω οι μεταφορέ, η γεωργία, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες αλλά και η αστυνομία, οι φορεί διαχείριση κρίσεων, η διαχείριση των συνόρων χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτά τα δορυφορικά συστήματα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να στηρίξουμε την πρόταση για το ευρωπαϊκό GNSS, γιατί έτσι οι ευρωπαίοι πολίτες θα υποφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που δίνουν αυτά τα συστήματα και θα έχουμε καλύτερη χρήση του Γαλιλαίου διαφυλάσσοντας και την εμπιστοσύνη του κοινού στα προγράμματα αυτά. Χαίρομαι για τη συμφωνία του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο που πέραν ε, του προϋπολογισμού προβλέπουν και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που κάνει σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του GNSS, ε, του, Ευρωπαϊκού, του Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό GNSS και της Υπηρεσίας του Διαστήματος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου για την διαμόρφωση ενός ανεξάρτητου αξιόπιστου συστήματος που προσφέρει έμπρακτες λύσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για την ασφάλεια στις μεταφορές, για την περιβαλλοντική προστασία και ούτω καθεξής. Επίση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που προσφέρουν τα συστήματα αυτά σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια πριν μεταφερθούμε σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Σα ευχαριστώ. Κυρία Τσικάου, δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ρούμπιχ. Κύριε Ρούμπιχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Τσικάου. Το ερώτημά μου είναι αν νομίζετε ότι το νέο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια για τα δεδομένα και την ασφάλεια δεδομένων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Λαμβάνοντας... Ότι τα συστήματα αυτά είναι ευρωπαϊκά πιστεύω ότι θα ε, συμμορφωθούμε το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, αυτά τα νέα ευρωπαϊκά συστήματα θα εξασφαλίσουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης ε, και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αντιλήσουν πολύ περισσότερα ωφέλη από το, από το σύστημα αυτό παρά από το GPS που εφαρμόζουν τώρα. Ο κύριος Ένι, ένα, ε, για... ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με το Καλιλαίο και το Έγνος επιτέλους το μονοπόλπο του βορειοαμερικανικού GPS που ελέγχει το πεντάγωνο θα σπάσει. Είναι καλό για την οικονομική, διπλωματική και πολιτική ανεξαρτησία των όλων της Ευρώπης. Είναι πολύ καλό νέο για την απασχόληση στην βιομηχανία, στις μεταφορές και στις ε, υπηρεσίες Ευρώπης. Φυσικά δεν θα γίνει εύκολα αυτή η κυοφορία. Ε, μπορούμε να επικρίνουμε την αρχική πολύ δαπανήρη κίνηση και την ε, εταιρική σχέση δημοσιοειδιωτικού φορέα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ε, η ευρωπαϊκή αυτή υποδομή παράγεται και χρηματοδοτείται από την Ένωση και είναι και ιδιοκτήτης ε, του συστήματο αυτού. Αυτό θα είναι υποφελές για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι μία από τα ελάχιστα σε ελάχιστε υπηρεσίε που είναι χρήσιμη, αποτελεσματική και στην υπηρεσία των πολιτών. Θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για όλες τις άλλες υπηρεσίες Επιτροπής, ε, αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εξυπηρετεί δυστυχώ μόνο τις χρηματαγορές. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Χίμπνερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Σήμερα Μιλάμε πραγματικά για ένα θέμα του 21ου αιώνα. Το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που θέλουμε να εφαρμόσουμε και ήδη χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη είναι από τα πιο σύγχρονα συστήματα που μας δίνει δυνατότητα πραγματικά ακριβούς πλοήγησης και μάλιστα εφαρμόζεται όχι μόνο ε, για τους, από τους οδηγούς, χρησιμοποιείται πάνω απ' όλα στην αεροπορία, στα σκάφη, στους ε, ψηφιακούς ταχογράφους, ε, στις ε, τράπεζες, ε, για αποστολές, courier. Ακόμη και από τους αθλητές χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα. Είναι ένα σύστημα πολύτως απαραίτητο. Και πραγματικά με το σύστημα αυτό μπαίνουμε στον 21ο αιώνα. Το έγνος είναι πολύ πιο προηγμένο τεχνολογικά σύστημα που χρησιμοποιείται από την πολιτική αεροπορία και από τις μεταφορές βιομηχανικών προϊόντων. Επίσης χρησιμοποιείται και από το στρατό. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι εμείς ε, στην Ευρώπη εφαρμόζουμε τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές και αξιοποιούμε πλήρως την τεχνολογία. Τα συστήματα αυτά βέβαια χαρίζουν ε, ανάπτυξη υποδομών στην Ευρώπη και φυσικά θα πρέπει να κατασκευάσουμε πολύ περισσότερους επίγειους σταθμού για να, ε, να καταργήσουμε αυτούς τους θύλακες που έχουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια για να επωφεληθούμε όλοι από αυτή τη τεχνολογία του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Στο Catch the Eye έχω έναν μόνο μιλητή, τον κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να δώσουμε πραγματικά μια ευκαιρία σε αυτήν τη νέα τεχνολογία που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και διότι ε, θα είναι προμηθευτές για το σύστημα και γιατί θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό αργότερα. Είναι μια νέα έννοια και γι' αυτό είναι ε, σημαντική ε, αυτή η έννοια της χρήσης του νέου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης γιατί θα μας δώσει και νέες εξαγωγικές δυνατότητες. Χρειαζόμαστε υψηλή τεχνολογία με υψηλά ποιοτικά κριτήρια. Συγχαίρω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή και ελπίζουμε ότι θα δώσει νέα πνοή στην ευρωπαϊκή οικονομία και βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ και θα ζητήσω από τον Επίτροπο να κάνει τις ε, τελικές παρατηρήσεις. Ο κ. Σταγιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες πληροφορίες για κάποια επιχειρήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η βιομηχανία διαστήματος αντιπροσωπεύει για την Ευρώπη ένα τομέα πολύ ποιοτικό, ένα τομέα που πρέπει πραγματικά να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες και είναι ε, τομέας κλειδί για την επανεκβιομηχανοποίηση της ε, Ευρώπης. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Ρούμπικ σε ό,τι αφορά την, το διεθνή χαρακτήρα που πρέπει να λάβουν οι, ε, οι επιχειρήσεις μας. Ειδικά στο τομέα του διαστήματος ε, ισχύει αυτό. Εγώ ε, πήγα σε μία αποστολή στο, στο Βιετνάμ, στην Βιερμανία κτλ. Ε, με αυτές τις χώρες θα προσυπογράψουμε πολλές συμφωνίες και πολλές από αυτές τις συμφωνίες αφορούν τον τομέα του διαστήματος. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλα όσα κάνει η Ευρώπη στον τομέα του διαστήματος από αυτές τις χώρες. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Γκάσπαρη, δηλαδή τι γίνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα σήματα του Γαλιλαίου να ε, μετατρέπονται σε υπηρεσίες. Σας ε, είπα ήδη ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για να δώσουν να, προσφέρουν υπηρεσίες αυτά τα σήματα του Γαλιλαίου και φέτος δύο φορές ήρθαμε σε επαφή με όλες τις βιομηχανίες, ενδιαφερόμενες βιομηχανίες του κλάδου, ε, βιομηχανίες που θέλουν να ε, εκμεταλλευτούν το Γαλιλαίο, μία φορά τον Ιανουάριο ε, στο Λονδίνο και μια δεύτερη φορά στο Φούκινο για να τεστάρουμε τα σήματα του Γαλιλαίου. Μιλάμε για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και τον επιχειρηματικό κόσμο, ούτως ώστε να πάρει ε, σάρκα και ωστά αυτή η νέα πραγματικότητα, τη χρήση δηλαδή των σημάτων αυτών σε διάφορους τομείς, προστασία ε, αστική, ε, αλληλεία, γεωργία, περιβάλλον, ενέργεια. Στη μία και 40 ενεργοποιήθηκε το σύστημα Κοπέρνικους για τις πλημμύρες όπως ας πούμε αυτή που έπληξε τη Σαρδινία με πολλούς θανάτους και μια καταστροφική κατάσταση. Το σύστημά μας ε, άρχισε να συνεργάζεται με τις Ιταλικές Αρχές λίγο μετά την α, πλημμύρα αυτή, μέσα στο το βράδυ εκείνο, μία και 40 όπως σας είπα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις καλές εγγύσεις που εξασφαλίζει το Γαλιλαίος είναι ένα σύστημα ευρωπαϊκό και η συνολική οργάνωση του συστήματος δίνει ε, περισσότερα εχέγγυα για την προστασία των δεδομένων. Πιστεύω λοιπόν ότι συνολικά το Γαλιλαίος αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόκληση, το είπε ο κύριος Νίμπλερ στα πλαίσια της παρέμβασής του. Ξεκινήσαμε πριν λίγα χρόνια, τώρα κάνουμε πολλά βήματα. Υπάρχει ε, το έγνος που είναι ήδη λειτουργικό και είναι ο πρόδρομος του Γαλιλαίου και που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το GPS, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερη ακρίβεια τα σήματα. Δουλεύουμε και για ένα άλλο project, το Κοπέρνικους. Θα ξεκινήσουμε σε κάνα δύο μήνες. Θα έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο στρατηγικών και πολιτικών διαστήματος και το Γαλιλαίος μόνο ένα τμήμα αυτών είναι. Ίσως το πιο φιλόδοξο, σύμφωνοι. Αλλά το Γαλιλαίο σε ορισμένου τομεί, κυρίω στην ε, πολιτική προστασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το Κοπέρνικου και να δημιουργήσει συνέργειε. δηλαδή τα σήματα του ενός συστήματος και τα σήματα του άλλου ε, συστήματος θα καταστήσουν πιο ασφαλή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε όμως να εξάγουμε κιόλα τη χρήση αυτών των σημάτων, των δικών μας ευρωπαϊκών συστημάτων, ώστε να βρούμε λύσει σε κρίσεις που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα, σε φυσικές καταστροφές. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η Ευρώπη είναι σκαπανέας εδώ. Και πριν ε, κλείσει τη δουλειά της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε έτοιμα τα, και λειτουργικά τα συστήματα του Γαλιλαίου. Ε, αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα που πετύχαμε και είναι σημαντικό ότι κερδίσανε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δείχνουν στους πολίτες ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο θυσίε, δεν είναι μόνο γραφειοκρατία, αλλά είναι και μία σειρά από αυτά αποτελέσματα προς το συμφέρον των πολιτών. Δίνουν περισσότερες ε, υπηρεσίες στους πολίτες ε, όλες αυτές τις προσπάθειες. Η Ευρώπη δίνει περισσότερες υπηρεσίες. Επίσης θα εξοικονομήσουμε τα επόμενα 20 χρόνια χρήματα χάρη στο Γαλιλαίος και τα υπολογίζουμε γύρω στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ξοδέψαμε 10 δισεκατομμύρια. Επομένω, θα έχουμε ένα θαυμάσιο ε, οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και πολιτικό και επιστημονικό και βιομηχανικό. Νομίζω λοιπόν ότι η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ σημαντική και ευχαριστώ ακόμα μια φορά τον κύριο Μαρινέσκο αλλά και όλους τους ευρωβουλευτές ε, που πάντα με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν αυτό το project και που δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει σε ορισμένου τομεί και να πετύχει ε, κάποια πράγματα. Ο τελευταίο μα ομιλητή στη συζήτηση είναι ο συγγητή μα, ο κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιος ρώτησε θα είναι αποδοτική επένδυση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συστήματα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ε, προσοδοφόρα αυτή η επένδυση. Και μάλιστα και εγώ προβληματίστηκα στις διαπραγματεύσεις ε, και είπα ότι θα είναι κρίμα να κατασκευάσουμε κάτι τόσο μακριά στο διάστημα που δεν θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχω πιστεί και το αντίθετο ότι θα ωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτε, γιατί θα αναπτύξουμε πολλέ εφαρμογέ χάρη στα συστήματα αυτά και με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια ε, για την ανάπτυξη των εφαρμογών. Επίση, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ε, να συνειδητοποιήσουν τα ωφέλη του Γαλιλαίου. Κάποιο ε, ρώτησε για την προστασία των δεδομένων. Το Γαλιλαίο έχει κρυπτογραφημένο σύστημα, κωδικοποιημένο, κάτι που εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αυτό είναι ο πρώτος κανονισμός που αφορά τον προπολογισμό του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και για το οποίο έχει εξασφαλιστεί συμφωνία. Και αυτό αυτή η συμφωνία οφείλεται στην αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους κοιόδης ηγητές αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την επικοδομητική συνεργασία. Επίσης να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία για τη συμβολή της στην συντόμευση των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλα στην εκπόνηση της έκθεσης. Και θα ήθελα να ευχηθώ εγκάρδια καλή επιτυχία στον Πίτρο Μποταγιάννη για να έχουμε μέχρι τα τέλη του 2014 ένα πραγματικά ποιοτικό σήμα. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο γύρω στι 12.30. Επόμενο θέμα της σημερινής διάταξη είναι η έκθεση κυρία Μπερέ, βασικά έγγραφα πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπερέ για 4 λεπτά.